Να σας καλωσορίσω όλους στη σημερινή συνεδρία της αντιπροσωπείας μας. Να καλωσορίσω επίσης όλους τους εκπροσώπους των διπλωματικών αποστολών, καθώς και τους εκπροσώπους Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, τον κύριο Πόνς, προϊστάμενο του Τμήματος για την Κεντρική Αμερική και το Μεξικό και την Καραϊβική. Η διαρμηνία θα παρέχεται στα ελληνικά, τα ισπανικά, τα πορτογαλικά και τα γαλλικά και η συνεδρίαση θα μεταδοθεί ζωντανά από την, μέσω του διαδικτύου. Ε, το σχέδιο της ημερήσιας διάταξης έχει διανεμηθεί σε όλους τους συναδέλφους, στα αγγλικά, στα ελληνικά και στα ισπανικά. Και αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, η, διά, η ημερήσια διάταξη θεωρείται ε, εγκεκριμένη. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι στις 9 Οκτωβρίου η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κούβα πραγματοποίησαν τον τέταρτο διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Αβάνα ήταν η πρώτη φορά που διεξήχθη επισήμω στο πλαίσιο τη Συμφωνία Ευρωπαϊκή Ένωση Κούβα για τον πολιτικό διάλογο και τη συνεργασία συμφωνία η οποία εφαρμόζεται προσωρινά από την 1η Νοεμβρίου του 2017. Ήταν επίση ο πρώτο από την σειρά πολιτικών διαλόγων που συμφωνήθηκαν κατά τη διάρκεια τη Συνόδου του Κοινού Συμβουλίου Ευρωπαϊκή Ένωση Κούβα, που στι 15 Μαου του 2018 η σχετική δήλωση επί του διαλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώματα τη ΥΠΑ τη εκπροσώπου τη Ευρωπαϊκή Ένωση για τα θέματα εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλεια κυρία Φεντερίκα Μογκερίνη βρίσκεται μέσα στον φάκελο που έχει ήδη διανεμηθεί. Και πάμε τώρα στο σημείο 3, που είναι η προετοιμασία τη επίσκεψη της αντιπροσωπείας μας στην Γουατεμάλα την 44η εβδομάδα του, του χρόνου, δηλαδή από τι 28 Οκτωβρίου και στην 1η Νοεμβρίου του 2018. Σήμερα η διάσκεψη των Προέδρων ενέκρινε την επίσκεψη της αντιπροσωπείας στη Γουατεμάλα για το χρονικό διάστημα που σας ανέφερα προηγουμένως. Ενέκρινε επίσης τη συμμετοχή στην επίσκεψη δύο επιπλέον μελών, ενός από την Επιτροπή της ΑΦΕΤ και ενός από την Επιτροπή της ΔΡΟΑ. Το σχέδιο του προγράμματος περιλαμβάνεται στους φακέλους και θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι εξακολουθεί να βρίσκεται σε σε αλλαγέ. Δηλαδή, όποιο έχει να προτείνει κάτι θα μπορούσε να περιληφθεί στι αλλαγέ που θα ήθελε. Κατά τη διάρκεια τη επίσκεψη, η αντιπροσωπεία θα συναντηθεί με εκπροσώπου των νομοθετικών οργάνων, τη κυβέρνηση, τη κοινωνία των πολιτών, των οργανώσεων των αυτόχθονων και του ιδιωτικού τομέα. Στόχο τη επίσκεψή μα, όπω πάντα, είναι να αποκομίσουμε μια ολοκληρωμένη και ισόρροπη εικόνα τη σημερινή πολιτική, οικονομική και κοινωνική κατάσταση στη Γουατεμάλα. Κύρια θέματα τη επίσκεψη είναι τα εξή η κατάσταση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων συμπεριλαμβανομένη τη περίπτωση τη κυρία Τσάβε, φιναλίστ του βραβείου Σαχάροβ για το 2017, η οποία αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη χώρα για λόγου ασφαλεία. Καταπολέμηση τη διαφθορά και στο πλαίσιο αυτό το μέλλον τη Διεθνού Επιτροπή κατά τη Ατιμορρησία του Γουατεμάλα. Διμερεί πολιτικέ και οικονομικέ σχέσει συμπεριλαμβανομένε τη εφαρμογή του εμπορικού πυλώνα τη Συμφωνία Σύνδεση Ευρωπαϊκή Ένωση Κεντρική Αμερική ασφάλεια και μετανάστευση, κοινωνικές και πολιτικές και μείωση της φτώχειας. Θα πραγματοποιηθεί επίση κοινή συνεδρία αντιπροσωπεία με το Παρλασέν, το οποίο θα αναδείξει το νέο του Προεδρείο, λίγο πριν από την επίσκεψη τη αντιπροσωπεία μα. Θα συζητήσουμε τρόπου για την ενίσχυση τη συνεργασία μα και για τον τρόπο με τον οποίο θα προχωρήσει η σύσταση κοινοβουλευτική κοινή κοινοβουλευτική επιτροπή Ευρωπαϊκή Ένωση Κεντρική Αμερική. Η αντιπροσωπεία θα ασκήσει επίση τα ελεκτικά τη καθήκοντα με την επίσκεψη ενό έργου που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Γουατεμάλα αυτή τη στιγμή εξετάζει ποιο είναι το καταλήτωρο έργο για την επίσκεψη. Επιπλέον, η αντιπροσωπεία θα εξετάσει διεξοδικά την εφαρμογή του εμπορικού πυλώνα τη συμφωνία σύνδεση με την Κεντρική Αμερική. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Πόνς, αναπληρωτή προϊστάμενο του Τμήματος για την Κεντρική Αμερική, το Μεξικό και την Καραϊβική της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και να ευχαριστήσω και την Επιτροπή σας, την αντιπροσωπεία σας για την πρόσκληση σήμερα θα μπορούσα να σας πω κάποια στοιχεία για το πώς βλέπουμε την υπόθεση στη Γουατεμάλα, να σας παρουσιάσω τις δράσεις τις οποίες έχει αναλάβει εκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, να αναφερθώ και στις διμερείς σχέσεις και είμαστε φυσικά στη διάθεσή σας για οποιοδήποτε άλλο θέμα θα μπορούσε να είναι σχετικό άλλωστε με την επίσκεψή σας και τις υπηρεσίες του Κοινοβουλίου έτσι ώστε να στεφθεί από επιτυχία η επίσκεψή σας. Ξέρετε ότι είναι περίπλοκη η συγκυρία στη Γουατεμάλα. Ξέρετε ότι στην ουσία είχε περάσει από μια σκληρή και πάρα πολύ συντριπτική θα έλεγα εμφύλια σύραξη η οποία ευτυχώς έχει μείνει πίσω μας τώρα αλλά είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί κανείς να αγνοήσει όταν προσπαθεί να αξιολογήσει την κατάσταση στη χώρα. Είναι μια πάρα πολύ πυκνοκατοικημένη χώρα της Κεντρικής Αμερικής, χαμηλού ως μέσου επίπεδου α, Ο πληθυσμός, ε, όπως είπα, αντιμετωπίζει προβλήματα φτώχειας. Υπάρχει φυσικά και ο ηθαγενής πληθυσμός, ο οποίος αντιμετωπίζει τα ίδια προβλήματα, αλλά σε ε, πιο σοβαρό επίπεδο από τους υπόλοιπους. Ε, τελευταίες οικονομικές επιδόσεις της χώρας είναι αρκετά ικανοποιητικές, ισχυρές θα έλεγα. Υπάρχουν όμως προβλήματα. Το αναγνωρίζει και η κυβέρνηση αυτή. Το θέμα της διαχείρισης των δημοσίου χρήματος, σαν παράδειγμα, έχει εν πολλής υπάρξει μια προσεκτική και επιφυλακτική διαχείριση των μακροοικονομικών δικτών, κάτι το οποίο δείχνει ίσως ότι οικονομικά η χώρα μπροστά της έχει ένα μέλλον αρκετά ικανοποιητικό. Να πω ότι έχει βέβαια δημιουργηθεί ένα θέμα τελευταία με την λεγόμενη Επιτροπή, Διεθνή Επιτροπή κατά της ατιμορρησίας στη Γουατεμάλα ο Επίτροπος Βελάσκες είχε να αντιμετωπίσει μια πολύ περίπλοκη κατάσταση και οδήγησε σε πολλά θετικά αποτελέσματα σε συνεργασία με την κυβέρνηση της Γουατεμάλα. Κανονικά, υπό συνθήκες, σε συνεργασία με τη Γενική Εισαγγελία της χώρας και όπως γνωρίζετε πρόσφατα, η συνεργασία αυτή πέρασε από πολύ δύσκολες στιγμές ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει εκφραστεί ξεκάθαρα και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς έχουμε επαναλάβει ε, την υποστήριξή μας στις εξαιρετικές εργασίες της ΣΥΣΥΓ, της ε, Διεθνούς Αυτής Επιτροπής, για την καταπολέμηση της διαφθοράς, να συνδυαστούμε με την κυβέρνηση της Γουατεμάλα, όπως το κάναμε στο παρελθόν, κάτι τέτοιο θα πρέπει να συνεχιστεί και στο μέλλον, να συνεχίσουμε λοιπόν την κοινή προσπάθεια σε συνεργασία με τη χώρα αυτή, έτσι ώστε τα πράγματα να εξελιχθούν με τον καλύτερο δυνατός, δυνατόν τρόπο. Φυσικά και σεβόμεθα πλήρως τις κυρίαρχες αποφάσεις του κράτους της Γουατεμάλα. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να ισχύει και για την Γουατεμάλα και με όλες τις χώρες με τις οποίες έχουμε σχέση. Ξέρετε ότι υπάρχει και μια ομάδα των 13 χωρών που είναι οι δωρήτριες χώρες και φυσικά εκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση παίζει σημαντικότατο ρόλο. Συμμετέχουν φυσικά και οι Ηνωμένε Πολιτείε και αυτό είναι κάτι το οποίο θα σας απασχολήσει και αυτό κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας. Ένα άλλο ίσως θέμα το οποίο μπορεί να σας απασχολήσει ε, στα πλαίσια των ε, είναι τα πλαίσια των προετοιμασιών για την εκλογική αναμέτρηση. Ξέρετε ότι θα γίνει προεδρική εκλογή τον μήνα Ιούνιο και τον μήνα Αύγουστο του 2019. μεσολαβεί περίπου κάτι παραπάνω από ένα χρόνο. συνεπώς ελπίζουμε οι διαδικασίες αυτές για την προετοιμασία των εκλογών να εξελιχθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και όπως πάντα η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι σε θέση να υποστηρίξει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις εκλογικές αυτές ε, προετοιμασίες. Και τέλος, ε, δεν θέλω να μακρηγορήσω, εσείς νομίζω ότι γνωρίζετε γενικά την κατάσταση στη χώρα της Γουατεμάλα, αλλά θα ήθελα ίσως να κάνω μια επιπλέον αναφορά στις σχέσεις τις οποίες έχουμε στα πλαίσια της συνεργασίας για την ανάπτυξη. Οι σχέσεις μας με τη Γουατεμάλα στον τομέα αυτό είναι σημαντικές. Έχουμε συνάψει με την Γουατεμάλα ένα πάρα πολύ σημαντικό α, πολιετές 750 εκατομμύρια σε τρεις τομείς για την περίοδο 14-20. Στο εσωτερικό του πολιετούς αυτού προγράμματος αντιμετωπίζονται θέματα όπως η διασφάλιση της προμήθειας τροφίμων, η επίλυση των συγκρούσεων, η ειρήνη, ασφάλεια και στήριξη για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομικής της χώρας. Κοιτάξτε, θα μπορούσαμε να αμακρηγορήσουμε σε σχέση με τις καλές σχέσεις που έχουμε με τη Γουατεμάλα. Έχουμε σταθερές σχέσεις με τη χώρα αυτή. Έχουμε καλές σχέσεις με την κυβέρνηση της χώρας. Έχουμε καλές σχέσεις με τον λαό της χώρας. Αλλά δεν έχω να πω κάτι άλλο. Απλά να πω ότι είναι απόλυτα διαθέσιμη η υπηρεσία εξωτερικών υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να συνεχίσει τη στήριξη ε, που παρέχει προς την Γουατεμάλα έτσι ώστε να ε, βοηθήσει στην ανάπτυξη της χώρας και να βοηθήσει και την καταπολέμηση του φαινομένου της ατιμορρησίας και του φαινομένου της ε, διαφθοράς. Δεν έχω κάτι άλλο. Αυτά αν θέλετε κάποια ερώτηση να κάνετε στη διάθεσή σας. Να σα ευχαριστήσω πολύ κύριε Πόντ και εγώ πραγματικά πιστεύω ότι αυτό το ταξίδι θα μα δώσει τη δυνατότητα να συγκεντρώσουμε σημαντικέ πληροφορίε για τη σχέση μα με την Γουατεμάλα. Ε, θα είναι πολύ σημαντικό για όλου του συναδέλφου που θα κάνουν αυτή την επίσκεψη. Δεν ξέρω αν ο κύριο ε, Αντιπρόεδρο θέλει να κάνει κάποια τοποθέτηση μετά από τις εξηγήσει τις οποίες μας έχει δώσει η Υπηρεσία Εξωτερικών Υποθέσεων και ο Φερνάντον Πόσο δεν έχουμε πάρα πολλά άλλα πράγματα να πούμε. Ε, εδώ και ένα περίπου χρόνο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε προετοιμάσει ένα ψήφισμα στο οποίο κάλυπτε όλα τα σημαντικά θέματα στα οποία αναφερθήκατε. Νομίζω λοιπόν ότι εξακολουθούν να ισχύουν όλα αυτά τα οποία είχαμε πει και θα πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειες τις οποίες από κοινού είχαμε ξεκινήσει. Ε, εμείς ε, είμαστε αρκετά ικανοποιημένοι ότι ε, τα προγράμματα στο πλαίσιο του ευρύτερου προγράμματος για την ανάπτυξη και τη συνεργασία προχωράει καλά. Υπάρχουν πολλά βέβαια τα οποία μένει να γίνουν ακόμα. Θα συνεχίσουμε να τα στηρίζουμε. Εγώ λυπάμαι για το συγκεκριμένο ταξίδι, δεν μπορώ να είμαι παρόν αλλά πέρασε αρκετός καιρός, ε, δεν είχε επιβεβαιωθεί το ταξίδι και δυστυχώς έπρεπε να πάω με μια αντιπροσωπεία της υποεπιτροπής αλληλείας στο Βιετνάμ. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η επίσκεψη την οποία θα κάνετε δεν είναι πάρα πολύ σημαντική και ενδιαφέρουσα. Και θα το συζητήσουμε Λοιπόν, δεν έχω κάτι άλλο να πω στη συγκεκριμένη περίπτωση. Θα συναντηθούμε λοιπόν ε, με τους συμμετέχοντες στο ταξίδι και θα κάνετε εξαιρετική δουλειά. Ευχαριστώ. Με δεδομένο ότι είναι δύσκολη μέρα σήμερα, οι συνάδελφοι δεν βρίσκονται στην αίθουσα εξαιτία του γεγονό ότι είναι και Πέμπτη, ταξιδεύουν αλλά και έχουν και άλλε επιτροπέ. Αυτό που θέλω εγώ να πω και να κλείσω την πιο μικρή επιτροπή που έχουμε κάνει μέχρι τώρα χρονικά είναι ότι περιμένουμε με ενδιαφέρον τι συμμετοχέ των συναδέλφων και φυσικά με ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον να ολοκληρώσουμε αυτό το ταξίδι και να επιστρέψουμε με τα συμπεράσματα, ούτω ώστε να τα συζητήσουμε στην Επιτροπή μα. Σα ευχαριστώ και πάλι για την παρουσία σα εδώ και για τον χρόνο που διαθέσατε. Είμαστε καλά. Μία ερώτηση θα είχα να θέσω στην προηγούμενη συνεδρίαση σε σχέση με το ταξίδι στην Κούβα, το οποίο για μια ακόμη φορά, εν πάση περιπτώσει, δεν θα γίνει. Είχαμε συζητήσει τα θέματα του διαλόγου Κούβα-Ευρωπαϊκή Ένωση και είχαμε πει ότι θα μπορούσαμε να στέλναμε μια επιστολή από πλευρά τη αντιπροσωπεία μα έτσι ώστε να μπορέσουμε, εν πάση περιπτώσει, να απευθύνουμε, να, να, να διαπιστώσουμε ότι δεν μας επιτρέπουν ουσιαστικά για μια ακόμη φορά. Η Κούβα κάνει ε, μια επιλογή στους προσκεκλημένους της. Όταν είναι ένας εκπρόσωπος κυβέρνησης ο οποίος είναι πολύ κοντά ε, στην κυβέρνηση της χώρας, ε, τον προσκαλούν χωρίς πρόβλημα. Λοιπόν, διαρωτώ με αν, έχει, αν δεν έχει αποσταλεί, να αποσταλεί μια επιστολή στην οποία να εκφράζουμε ε, την, ε, την άποψή μας και να μας δώσετε και αντίγραφο αν γίνεται. Όχι, δεν έχει σταλεί κάποια επιστολή τέτοια. Βρίσκονται εκείνοι μα απαντήσουν ότι βρίσκονται ε, στη διαδικασία αναθεώρηση του συντάγματο, αλλά είναι κάτι που μπορεί να γίνει, δεν είναι κάτι που θα το αποφύγουμε. Δεν υπάρχει λόγο δηλαδή. No, perdón, presidenta, pero, pero la carta no tiene nada que Κοιτάξτε, η επιστολή μας αυτή δεν πρέπει να έχει καμία σχέση μετά τη συνταγματική αναθεώρηση. Να πούμε ότι λυπούμεθα γιατί για μια ακόμη φορά δεν μας επετράπει, δεν επετράπει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να κάνει μια επίσημη επίσκεψη. Αυτό μόνο. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το συμβατό ε, και με αυτά τα οποία έχουμε συζητήσει στα πλαίσια και του ΜΕΚΟΣΑ. Αντιπρόεδρο, είστε μαζί, θα την κάνουμε την επιστολή. Δεν είναι κάτι που θα κάνω και δεν θα το ξέρετε, Θεού. Ε, είναι κάτι που θα το συζητήσουμε. Ο τρόπο που θα ε, συνταχθεί αυτή η επιστολή είναι κάτι που θα κοινοποιηθεί και θα μαζί θα το ολοκληρώσουμε. Ευχαριστώ.